προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αφορά την αυτόνομη οδήγηση. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο συντάκτης της ερωτήσεως, ο κύριος Ερτούγ. Ποιος είναι ο κύριος Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. με καλά πιστεύω που φέραμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Γιατί είναι σημαντικό και για το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Ένωση και για τις τεχνικές, τεχνολογικές εξέλιξεις. Ο τομέα, ο κλάδο αυτοκινητοβιομηχανία, αγαπητοί συνάδελφοι, βρίσκεται σήμερα στάδιο ταχεία ανάπτυξη. Ενώ κατά τα τελευταία δέκα έτη ορισμένα συστήματα υποβοήθηση του οδηγού έχουν σταδιακά εφαρμοστεί και βελτιστοποιηθεί η εν μέρη αυτόνομη οδήγηση είναι περίπου έτοιμη να τεθεί σε ισχύ και πρόκειται για το επόμενο βήμα. Το 2016 τα πρώτα μοντέλα αυτοκινήτων που είναι εξοπλισμένα με συστήματα εν μέρη αυτόνομη οδήγηση όπω πλήρη δυνατότητα αυτοδύναμου παρκαρίσματο, αποφυγή κυκλοφοριακή συμφόρηση κτλ. θα εισαχθούν στην αγορά. Η πρώτη γενεά των πλήρω αυτόνομων οχημάτων βρίσκεται επί του παρόντο υπό ανάπτυξη από του κατασκευαστέ οχημάτων και του μηχανικού συστημάτων με γενικότερο στόχο τη αγωγή του στην αγορά το 2030. Εν ώψη αυτών των ταχύων. εξελίξεων, το τομέα μεταφορών τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει επιγόντω να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, να παραμείνει ανταγωνιστικό εναντί άλλων περιφερειών κτλ. Και έτσι το δυναμικό τη αυτόνομη οδήγηση δεν αφορά μόνο τον τομέα των μεταφορών. Μπορεί να οδηγήσει σε ταχύτατε εξελίξει και σε άλλου κλάδου. επιμελητία, γεωργία, ορυχία, στην, ε, στη χωροταξία επίσης ε, των αστικών κέντρων και ε, τη διαμόρφωση συνθήκων οδήγησης. Θα χρειαστούν νέες, νέα μέτρα. Υπάρχουν ανάγκες για διαφορετικές δοκιμές και διαδικασίες ελέγχου. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ωστόσο, δεν υπάρχουν συγκεκριμένες στρατηγικές ορατές τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής για το πώς θα αντιμετωπιστεί η αυτόνομη οδήγηση. Πάντως υπάρχει μια σειρά βασικών διαδικασιών ελέγχου και δοκιμών που πρέπει εξαπαντούς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστεί όχι μόνο για να έχουμε αποτελεσματική και ασφαλή ε, αποτελεσματικό και ασφαλή τομέα των μεταφορών, αλλά και για να δώσουμε σαφείς οδηγίες και κατευθυντικές γραμμές στην ε, αυτοκινητοβιομηχανία μας και βέβαια να τη βοηθήσουμε στη συνεργασία και με άλλες μεγάλες αντίστοιχες περιφέρειες οικονομικές όπως οι ΗΠΑ για ε, συνεργασία και σε τεχνικού όρου. Πρέπει τα αισθήματα αυτά λοιπόν να απασχολήσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δώσει ε, πιστικέ και μακροπρόθεσμε απαντήσει. Και εδώ έχουμε το ζήτημα τη ευθύνη, τη αστική ευθύνη. Όταν λοιπόν αφαιρείται από τον έλεγχο του οδηγού ε, η καθοδήγηση του αυτοκινήτου, την αστική ευθύνη ποιος την αναλαμβάνει. Έχει απασχολήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ζήτημα τη προσαρμογής ε, των σχετικών διατάξεων περί αστική ευθύνη. Ερωτηματικό. Επίσης, σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την κυβερνό ασφάλεια. Επικοινωνία μεταξύ οχημάτων, αλλά και μεταξύ οχημάτων και υποδομών, που πρέπει να γίνεται με τρόπο ασφαλή και απρόσκοπτο με σεβασμό βέβαια των προσωπικών δεδομένων, τα δεδομένα των οχημάτων και δι των πολιτών της Ευρώπης. Πώς σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα προστατέψει στην επικοινωνία με τις δομές αυτές. Υπάρχουν ζητήματα εκκρεμίως προς τις υποδομές επίσης. Τα, αυτόματα, τα αυτόνομα οχήματα μπορούν να ενταχθούν στις υποδομές όπως αυτές έχουν τώρα, οδικές υποδομές και άλλες ή χρειάζονται κάποιες προσαρμογές και τότε ποιος θα τις χρηματοδοτήσει τις προσαρμογές αυτές. Και ως προς τις εγκρίσεις τύπου ερωτηματικά υπάρχουν επίσης πολλά. Τα αυτόνομα οχήματα, κυρία Επίτροπε, χρειάζονται διαφορετικές δοκιμές και διαδικασίες ελέγχου και θα πρέπει να προσαρμοστεί η φυστάμενη νομοθεσία για την έγκριση τύπου οχημάτων. Έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μελετήσει με βάση παραδείγμα του κανονισμού Οικονομικής Επιτροπής των ΗΠΑ για την Ευρώπη, της ΟΝΕΣΕ, μια τέτοια εξέλιξη δεδομένων των πολλών ζητημάτων και ερωτημάτων που τίθενται λοιπόν και που απασχολούν και τους συναδέλφους, θέλω να ρωτήσω εάν έχει αρχίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονεί μια στρατηγική για την αυτόνομη οδήγηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αν συμφωνείτε κύριε Επίτροπε ότι υπό το φως της αυξανόμενης σημασίας της αυτόνομης οδήγησης είναι απαραίτητη η έγκαιρη δημοσίευση μιας πράσινης βίβλου. Και σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε κύριε Ερτούγκ. Και τώρα η κυρία Τάισεν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, αυτού του είδους υποβοήθηση του οδηγού βοηθά την ασφάλεια, τη ροή της κυκλοφορίας, είναι κάτι πιο αποτελεσματικό και πιο φιλικό στο περιβάλλον. Χρειάζεται να υπάρχει περισσότερη συνέργεια και πιο στενή συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε την δήλωση του Άμστερνταμ που σήμερα εγκρίθηκε στα πλαίσια του άτυπου Συμβουλίου Μεταφορών. Επ' αυτού είναι ξεκάθαρη αυτή η δήλωση, η διακήρυξη και επομένω είναι η αρχή μιας ε, ευρωπαϊκής στρατηγικής όσον αφορά την αυτόνομη οδήγηση. Σήμερα επομένω συζητήθηκαν αυτά και γι' αυτό το λόγο και ο συνάδελφο Μπούλιτ δεν είναι εδώ. Έπρεπε να παραστεί εκεί και άρα θα σα τα πω εγώ σήμερα. Εμεί έχουμε ξεκινήσει διάλογο με τα κράτη-μέλη, τι κρατικέ αρχέ και τον ιδιωτικό τομέα, το ώστε να υπάρχουν συστήματα ε, και μια ολόκληρη πλατφόρμα όσον αφορά τα αυτόνομα οχήματα. Στόχος είναι το 2030. Τότε θα βγουν στην παραγωγή τα οχήματα αυτά, όπως έχει πει και ο Επίτροπος και είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε μια τέτοια ευρωπαϊκή στρατηγική και αυτό θα πλαισιωθεί από έρευνα, και καινοτομία, την αντίστοιχη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα και η μία εδώ είναι ο στόχος. Επομένως αυτή η τεχνολογία για τα αυτόνομα οχήματα είναι μια τεχνολογία που εξελίσσεται γρήγορα. Έχουμε αυτά τα πολύπλοκα συστήματα και στόχος είναι η περισσότερη ασφάλεια αλλά και άνεση στην οδήγηση. Ε, υπάρχουν κάποια τέτοια συστήματα ε, μερικής ε, αυτονομίας και θα προβούν στην πλήρη αυτονομία στο μέλλον. Όμως θα πρέπει πάνω απ' όλα να πρετανεύει η ασφάλεια και η διαδικασία προς την αυτονομία θα πρέπει να οδηγεί σε περισσότερη ασφάλεια και θα πρέπει να αποκλείει κάποιους κινδύνους, μην προσθέτει κι άλλους. Στην ερώτησή σας αναφέρεστε σε αυτές τις προκλήσεις της ε, αυτονομίας των οχημάτων. Έχουμε ένα νομικό πλαίσιο θα πρέπει ομένως στο πλαίσιο αυτό που αφορά την οδήγηση να προσαρμοστεί στα αυτόνομα οχήματα και να ε, διέπονται από αυτό το νομοθέτημα όλοι οι χρήστες των δρόμων να εφαρμοστούν οι διεθνείς ε, συμβάσεις ιδίω όσο πρέπει να ισχύσει να ληφθεί η σύμβαση της Βιέννης για την οδική κυκλοφορία και φυσικά οι οδικοί κώδικες. Οπότε έχουμε η στην την προσπάθεια και κινούμε θα σε διεθνές επίπεδο. Άρα θέλουμε να έχουμε όσο γίνεται μεγαλύτερη ε, ασφάλεια σε επικοινωνία αλλά και στην προστασία ιδιωτικότητας και προσωπικών δεδομένων. Ε, αυτά όλα θα πρέπει να τα συνειδητοποιήσει και ο κόσμος και θα πρέπει επομένως να κινηθούμε και με τη στρατηγική ε, για τα ψηφιακά έχουμε τον νέο κρονισμό για την προστασία των δεδομένων. Οπότε να υπάρχει ε, ενιαία νομοθεσία κοινωτικό δίκαιο για την προστασία των δεδομένων. Αλλά αυτά τα εξετάσουμε και στα πλαίσια της πλατφόρμας που θέλουμε να ισχύσει. Έχουμε επομένω την πρωτοβουλία για το 2030 όσον αφορά τα πάρα πολύ αυτόνομα οχήματα και θέλουμε τώρα να δούμε τι θα αλλάξει και αν θα αλλάξει κάτι όσον αφορά τα επίπεδα της αυτονομίας. Επίσης έχουμε το θέμα της ε, κατασκευής δρόμων που θα πρέπει να προσαρμοστεί στη νέα τεχνολογία. Ε, αυτή η πλατφόρμα που ασχολείται με την αυτονομία τα έχει λάβει αυτά και καλύπτονται όλα τα ζητήματα αυτά από την πρωτοβουλία για το 2030 επίσης να αναβαθμίσουμε τα δίκτυα επικοινωνιών και αυτά συζητούνται στην ε, Στρογγυλή Τράπεζα Υψηλού Επιπέδου για την αυτόνομη ε, οδήγηση. Τώρα, όσον αφορά τις ε, δοκιμές, επιθεωρήσεις, ελέγχους και την έγκριση τύπου. Αυτά τα πάρα πολύ αυτόνομα οχήματα θα πρέπει να κληρούν όσα ισχύουν ε, ήδη ας πούμε για τις εκπομπές και οι επαφές συνεχίζουν σε επίπεδο UNESE, Επιτροπή Ηνωμένων Εθνών, ώστε να προσαρμοστούν όλοι οι κανόνες σε αυτές τις εξελίξεις. Και σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε. Τώρα θα ακούσουμε του εκπροσώπου των πολιτικών ομάδων εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, κατά παράδοση. Ο κύριος Πόλτσακ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δυστυχώς, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και έχει μπει τελευταία στην ημερήσια διάταξη της Πέμπτης, αλλά πρέπει να αρχίσουμε να το συνηθίζουμε πια. Θεωρώ δε πονίδιστο το ίδιο ότι η ομάδα της Μαρίν Λεπέν και άλλων και άλλοι ευρωσκεπτικιστές δεν είναι εδώ όταν συζητούμε θέματα σοβαρά όπως η μετανάστευση. Μπορώ να συμφωνήσω λοιπόν εν πολύ στα όσα είπε ο κύριος Ερτού, συντάκτης της ε, προφορικής ερώτησης. Όντως ο κλάδος της, αυ της αυτοκινητοβιομηχανίας βρίσκεται σε, μια, σε ένα σημείο καμπής, σαν να περνάμε από το αερόστατο στο αεροπλάνο. Ήδη γίνονται δοκιμές στην πρώτη γενιά αυτόνομων οχημάτων. Και θα τα δούμε να κυκλοφορούν στους δρόμους μας τα επόμενα χρόνια. Πρόκειται για ιστορική περίοδο. Πάντως με βάση τα τελευταία δεδομένα δεν θα είναι τόσο πρόσκοπτη αυτή η οδήγηση. Με βάση πρόσφατες πληροφορίες, στατιστικές από την Καλιφόρνια των ΗΠΑ, μία από τις λίγες ε, πολιτείες ανά τον κόσμο που επιτρέπουν την χρήση αυτόνομης οδήγησης ε, στο... στους δρόμους της έχουν καταγραφεί μέσα σε ένα χρόνο πάνω από 3.000 προβλήματα. Η Mercedes-Benz συγκεκριμένα 1.051 επεισόδια ε, δυσλειτουργίας με δύο μόνο οχήματα στην πολιτεία της Καλιφόρνιας της Mercedes-Benz στην περίοδο αυτή 1051 περιπτώσεις προβλημάτων και δυσλειτουργιών. Πρέπει λοιπόν να θυμάμαστε ότι όρος ο κάνει φαίνει η ασφάλεια στις οδικές μεταφορές. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποφεύγονται πάντοτε ή αδίποτε ατυχήματα. Πρέπει λοιπόν να δούμε αυτό το ζήτημα, ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε 100% τα ατυχήματα. Και τότε να περάσουμε στο επόμενο ερώτημα, ποιο θα έχει την αστική ευθύνη σε περίπτωση ατυχημάτων. Επαναλαμβάνω λοιπόν την ερώτηση. Πώ θα προσαρμοστεί το ισχύον νομικό πλαίσιο. Σκοπεύει να τροποποιήσει την ε, συνθήκη της Βιέρης του 1968 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε αυτό πρώτα. Και ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πόλτσακ. Εκ μέρους των σοσιαλιστών τώρα το λόγο έχει η κυρία Ινές Αγιάλα Σέντερ. μισή λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ για τη γενοδορία. Λοιπόν, ο κλάδος αυτοκινητοβιομηχανίας φυσικά και θέλει να προχωρήσει γρήγορα με οχήματα από το δίζελ και τη βενζίνη με οδηγούς. Τώρα βρισκόμαστε στον κόσμο της ψηφιοποίησης και των ρομπότ που σιγά σιγά θέλουν να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους. Υπάρχουν και κίνδυνοι. Τον οδηγάει κανείς, πιστεύω, ότι προς το παρόν δημιουργεί αίσθηση και σε πολλούς αρέσει. Η σημερινή ασφάλεια έχει σαν αποτέλεσμα ε, μερικές φορές να λέμε ότι δεν φταίει ο οδηγός, αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό. Στα αεροπλάνα έχει συμβεί, έχουν αυτοματοποιηθεί τα αεροπλάνα και όταν βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης, οι πιλότοι δεν καταφέρουν να πάρουν ε, τα ενία και τον έλεγχο του αεροπλάνου, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η αυτοματοποίηση που την έχουν κάνει οι άνθρωποι, φυσικά δεν την έχει κάνει κανένας ε, η Περγίνος. Συνεπώς, νομίζω ότι δεν ε, πρέπει να μας ε, διέπει ένας υπερβολικός, μια υπερβολική αισιοδοξία και φιλοδοξία με αποτέλεσμα να γνωρούμε τους πραγματικούς κινδύνους. Λοιπόν, είτε πρόκειται για οδηγού, είτε για οδηγού φορτηγών, είτε τρένων, είτε οτιδήποτε, Ας κοιτάξουμε πρώτα τη μείωση των κοινωνικών δικαιωμάτων όλων αυτών και να προχωράμε πάρα πολύ προσεκτικά. Και αν δεν οδηγούμε εμεί τελικά τα οχήματα ή θα τα οδηγούμε από απόσταση με τηλεκατεύθυνση, γιατί εντάξει και αυτό είναι οδήγηση αλλά είναι από μακριά. Το θέμα είναι να δούμε ποιοι κίνδυνοι ελοχεύουν κάθε φορά και ποιο είναι το νομικό πλαίσιο. Η μηχανική θα προχωρήσουν σε αυτήν την αυτόματη οδήγηση, χωρίς όμως να έχουμε αντιμετωπίσει άλλα προβλήματα, όπως είναι η ρήπανση από τα οχήματα. Ίσως αυτό πρέπει να κοιτάξουμε πρώτα. Και για τα φορτηγά, όπως λέει και η Επίτροπος, θα ήθελα να επενθυμίσω ότι τελικά καταλήγουμε να αντικαθιστούμε το τρένο από τους δρόμους και όχι το αντίθετο. Θέλουμε ναι. να εναρμονίσουμε τους κανόνες, γι' αυτό πιστεύω ότι στην περίπτωση των αυτοματοποιημένων οχημάτων θα πρέπει να είμαστε σε θέση να έχουμε ένα νομικό συνενετικό πλαίσιο πριν να αρχίσουμε ο καθένας από τη δικιά του την πλευρά να φτιάχνει αυτό που θέλει, γιατί αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχουν διάφορα πειραματικά σχέδια που γίνονται, που όμως μεταξύ τους δεν είναι διαλειτουργικά. Στηρίζω λοιπόν τον κύριο Ερτούκ για το ότι επήγει να έχουμε μια λευκή βίβλο όπου όλες αυτές οι πτυχές θα αναφέρονται για να μην έχουμε κατακαιρματισμό και έλλειψη συνοχής με κοινωνικές επιπτώσεις. Τα κοινωνικά δικαιώματα. Το κόστος των υποδομών, οικονομικές επιπτώσεις πρέπει να μετρεθούν πάρα πολύ καλά πριν αρχίσουμε να σκεφτόμαστε ότι θα καταλήξουμε στο αυτοκινητάκι μας να καθόμαστε και να διαβάζουμε ή να παίζουμε ενώ μας πηγαίνει το αυτοκίνητο από μόνο του όπως γίνεται με τα τρένα περίπου σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα για την Ίσια, κυρίως Ζλωτόφσκι. Βλέπω ότι παγίω σήμερα μιλάτε για την πολιτική σώμα. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Λοτόφ και κυρίε και κύριοι. Το μέλλον των μεταφορών είναι κάτι για το οποίο θα πρέπει τώρα να μας προγραμματίσει διότι κάθε μέρα κατεβάζουμε καινούργιες ιδέες, καινούργιες ε, φρέσκες καινοτομίες τέλος πάντων για ε, κάποιες υποδομές που βέβαια ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί διότι τα το γίνεται δεν είναι απλά μια ιδέα. Ε, μια ιδέα, συγγνώμη, είναι κάτι το οποίο ήδη το έχουμε πραγματοποιήσει και έχει μπει στο δρόμο του από τους κατασκευαστές που και μια επανάσταση που θα λύσει πολλά από τα σημερινά προβλήματα κινητικότητας περιβάλλοντος αλλά και ασφάλειας θα έχουμε επομένω αυτά τα ευφύ αυτόνομα αυτοκίνητα. Αυτό πάει να πει καλύτερη ροή της κυκλοφορίας με λιγότερα ε, ατυχήματα, καλύτερη αξιοποίηση των πόρων και ακριβώ όπω την περσμένη εβδομάδα, αυτό θα είναι μια επανάσταση και για την οδική μεταφορά. Όμω θα πρέπει πάσα αλλαγή να περνάει από πολύ σωστή προπαρασκευή, γιατί είναι και το θέμα του τι θα γίνει από πλευρά αγορά-εργασία. Άρα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει την αναγκαία ανάλυση για την ευρεία χρήση τέτοιων αυτοκινήτων και σα ευχαριστώ. Εγώ σα ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος, πολύ σημαντικά τα όσα μα είπατε και τώρα η κυρία Χαράντσοβα. Για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ακούσαμε για όλα αυτά τα θαύματα που θα φέρει στη ζωή μας η αυτόνομη οδήγηση, η αυτόνομη ε, ε, ε, αυτοκίνητο. Εγώ περιμένω πώς και πώς να έχω τέτοιο συνδεδεμένο αυτοκίνητο και βέβαια όλος αυτός ο ενθουσιασμός δεν απαντά όλα μας τα ερωτήματα. Πώς θα προσαρμοστεί σε αυτά τα πράγματα τα καινούργια η βιομηχανία, πώς θα εξασφαλίσουμε την ασφάλεια, πώς θα εξασφαλιστούμε από τις κυβερνοεπιθέσεις, τι θα γίνει με τα δικαιώματα των καταναλωτών, πώς θα προστατευτούν τα δεδομένα, τι θα γίνει με την αστική ευθύνη. Είναι τόσο περίπλοκα τα ζητήματα που δεν μπορεί ένας μόνο να τα απαντήσει γιατί θα πρέπει η βιομηχανία να εμπλακεί στην προβληματική και θα πρέπει να έχουμε ένα εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο το οποίο να είναι ευρύτερο από τα θέματα τα τεχνολογικά. Άρα θα πρέπει να συνεργαστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Η ίδια δε η βιομηχανία μας θα πρέπει να κάτσει και να δει πώ θα λάβει υπόψη την ασφάλεια τα δεδομένα, το τι θα γίνει με τη διαχείριση των δρόμων, καινούργια μοντέλα επιχειρηματικά. Άρα βλέπουμε ότι θα πρέπει να πάρα πολλέ ε, ε, αλλαγέ και θα πρέπει να γίνει ταχεία προσαρμογή. Ιδάλω καμία εταιρεία στην Ευρώπη, καμία αυτοκινητοβιομηχανία ε, δεν ε, πρόκειται να τα πάει καλά. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη και στην επιχειρηματικότητα και αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα αξιοποιήσουμε την τεχνολογία ε, και την εμπειρία των πολιτών και για πώς προσθέτουν τις ζωές και για όλους αυτούς τους λόγους θα πρέπει να γίνει η ασφάλεια μεγαλύτερη και προς τα εκεί πρέπει να πάμε εδώ και τώρα. Σε ευχαριστούμε πολύ λέει ο Πρόεδρος. Για τους πρασίνους τώρα. Η κυρία Καρίμα Ντελή. Έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε το συνδεδεμένο αυτοκίνητο και το αυτόνομο. Σε 10 χρόνια θα το έχουμε και αυτό. Είναι μια μικρή επανάσταση που απαιτεί επαναστατικές αλλαγές. Γιατί εδώ, στο ημικύκλιο, αυτό που κάνουμε είναι ότι εκπονούμε το δίκαιο του ρομπότ. Όντω λοιπόν χρειάζεται νομοθεσία. Αν υπάρχει ατύχημα, ποιο θα είναι υπεύθυνο, μια που δεν θα είναι πια ε, ο οδηγό, θα είναι ο κατασκευαστή, αυτοί που το κατευθύνουν, αυτοί που φτιάχνουν τι κατάλληλε εφαρμογέ στο διαδίκτυο. Πρέπει να φροντίσουμε όλε οι προδιαγραφέ να τηρούνται. Και οι σχολέ ε, οδήγηση θα είναι περίτε. Τώρα χρειαζόμαστε ένα πραγματικό κώδικα υπέρ της οδικής ασφάλειας, αλλά και διαφάνεια ώστε και οι επιβάτες αλλά και οι εργαζόμενοι να μην είναι θύματα του ανταγωνισμού. Γιατί το βλέπουμε ότι σήμερα κανένας κατασκευαστής δεν σέβεται τις προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο επιβάτης όμως τελικά την πληρώνει. Το βλέπουμε και στη Γαλλία και στο Βέλγιο με το σκάνδαλο της Volkswagen που ερευνά το κοινοβούλιο μας. Οπότε το λέω, στην ε, ανακοίνωσή σας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάτε για διεθνή συνεργασία μεταξύ των κατασκευαστών. Εγώ λέω ότι χρειάζεται μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποίησης για τον αυτοματισμό αυτό. Και βέβαια, με τι θα κυκλοφορούν τα οχήματα αυτά, με τι καύσιμα θα δώσουμε μια δεύτερη γενιά, δεύτερη ευκαιρία στο ντίζελ. Όχι, τη στιγμή που προκαλεί καρκίνο. Άλλη μια απάτη λοιπόν για τους καταναλωτές. Πρέπει να φτιάξουμε ένα αυτοκίνητο το οποίο θα ρηπαίνει πολύ λιγότερο. Αν το αυτόματο όχημα ε, ενισχύει τον ανταγωνισμό και μειώνει τις άλλες μορφές μεταφορών, και σκέφτεται περισσότερο τον ανταγωνισμό παρά της πόλης ή τον άνθρωπο, ε όχι. Τη βιώσιμη ε, κυκλοφορία και μεταφορά πρέπει να σκεφτόμαστε και υπάρχουν και άλλες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πότε θα, θα αποφασίσουν οι χώρες να κάνουν διαβουλεύσεις με τους καταναλωτές, με την τοπική αυτοδίκηση και την χωροταξία πρέπει να την ξαναδούμε. Τα οχήματα αυτά θα προστατεύουν τα δεδομένα. Και τι θα γίνει με τα εκατομμύρια εργαζόμενους σήμερα στις μεταφορές που είναι οδηγοί δηλαδή και που ξαφνικά θα βρεθούν χωρίς δουλειά. Οι νομοθέτες δεν ξέρουν τι να κάνουν σε αυτή τη διαμάχη μεταξύ των ε, οδηγών ταξί και των Uber. Τι θα κάνουν λοιπόν σε αυτή την περίπτωση. Και ολοκληρώνω πρόεδρε. Το αυτοκίνητο κάνει την επανάστασή του. Εντάξει, τη χρειαζόμαστε. Αλλά ας μάθουμε και από τα σφάλματα των κατασκευαστών του παρελθόντος. Δεν θα λειτουργήσει καμία τεχνολογία αν από πίσω δεν υπάρχουν ευφύς άνθρωποι. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Να τηρείτε το χρόνο σας παρακαλώ. Τώρα, συνεχίζουμε και περνάμε στους άλλους ομιλητές. Κύριος Λάμπερτ Κόχ πρώτα. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι βεβαίω που μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα της ε, αυτόνομης οδήγησης ε, σε τόσο πρώιμο στάδιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει το δεύτερο στάδιο που είναι η ψηφιοποίηση και η βιομηχανία 4.0. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο στις εξελίξεις τεχνολογικές που θα μπορούσε να αλλάξει μεταφορές μας ε, σε τέτοιο βαθμό. Από την αυτόνομη οδήγηση θα περάσουμε και στην οδήγηση χωρίς οδηγό. Θα χρειαστεί όμως αλλαγή και προσαρμογή του νομικού πλαισίου. Τα αυτόνομα αυτοκίνητα μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες κυκλοφορίας στους δρόμους, γιατί στα οχήματα με κινητήρα το συντριπτικό ποσοστό των ατυχημάτων οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος, αλλά μπορούν να μειώσουν και ε, την κατανάλωση καυσίμων και την ε, ώρες αυτοκινήτων προς εκ τούτου τα μποτιλιαρίσματα στους δρόμους οι δοκιμέ πρέπει να προχωρήσουν. Πρέπει να προχωρήσουν και με του αυτοκινητοδρόμου τη Γερμανία, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε και σε θέματα προστασία των προσωπικών δεδομένων ε, πώ μπορούμε να προστατευτούμε, πώ μπορούμε να προστατεύσουμε τα δεδομένα από του hacker, αλλά και ταυτόχρονα πώ μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα δεδομένα για να γίνεται σωστή επικοινωνία. Και αν τελικά φτάσουμε στην σύγκρουση, στο τρακάρισμα, τι θα συμβαίνει, γιατί το θέμα δεν είναι μόνο... Ε, οικονομικό, είναι και ηθικό. Θα καλείται ένα αυτοκίνητο μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου να λάβει την απόφαση εάν θα στραφεί για να πέσει πάνω σε ένα κορμό δέντρου ή εάν θα χτυπήσει ένα πεζό. Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με τον 21ο αιώνα και την οδήγηση που θα ταιριάζει σε αυτή την περίοδο. Ευχαριστώ πολύ. Μα με κίνησε ένα, μισή λεπτό. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, όποιος έχει δει το Star Trek έχει διαβάσει Καζιμιστέλη θα ξέρει ότι αυτά τα οράματα τα είχε ο άνθρωπος από πολλά χρόνια για την αυτόνομη οδήγηση. Ένα από τα κύρια ζητήματα βεβαίως που τίθενται είναι η ασφάλεια. Πρέπει να υπάρχουν πολλοί προηγμένα συστήματα ε, τεχνολογικής καθοδήγησης και δυνατότητες πρόληψης. Βεβαίως οι διαδικασίες των δοκιμών θα είναι τελείως διαφορετικές από αυτές των παραδοσιακών οχημάτων και θα έχουν αυτές τεράστια σημασία. Ένα άλλο ζήτημα είναι η ασφάλεια. Δεν θέλει κανείς να πέσει θύμα απαγωγής την ώρα που έχει βγει για να αλλάξει τον τροχό του αυτοκινήτου του. Χρειάζεται μια καλή στρατηγική για τον τομέα αυτό των μεταφορών και δεν πρέπει να λησμονούμε το Skynet, τη μεγάλη αυτή αμοιβαία ευθεία που θα επιτρέψει κάποια μέρα στα ρομπότ να έχουν αυτόνομη σκέψη και βούληση. Και ίσως κάποια ώρα έρθει η στιγμή και εμείς να διερωτηθούμε εάν έχουμε τον έλεγχο της ίδιας μας της ζωής. Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, Μπιλουά Μπαραντίκα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε και κύριε Επιτροπή. Και πάλι, νομίζω ότι η πρόοδος της τεχνολογίας όσον αφορά την αυτόνομη οδήγηση τώρα δημιουργεί ένα σωρό ζητήματα θεσμικά και νομικά τα οποία θα πρέπει με συνέπεια και συνολικά να αντιμετωπίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την ε, νομοθεσία και συγκεκριμένα την στρατηγική για τις κρατικές επενδύσεις. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά για έχουμε την συνδεσιμότητα μεταξύ των ε, οχημάτων και των ε, υποδομών για τα οχήματα. Και εδώ έχει σημασία η βριζοζωνικότητα, έχουμε τον Γαλιλαίο, αλλά δυστυχώς εκεί έχουμε καθυστερήσεις και περικοπές. Για τι θα κάνετε όσον αφορά τι επενδύσει κύριε Επιτρόπο του ώστε αυτά τα οχήματα να μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί θα ήταν θλιβερό κάποια προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με αθέτηση υποχρεώσεων επενδυτικών σε κάποια κράτη-μέλη να μην μα αφήνουν να εκμεταλλευτούμε αυτά τα οχήματα. Επίση, θα θέλω να μου πείτε κατά πόσο τώρα θα αναθεωρήσετε τα των ε, πανευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Τέλος, τα χαρακτηριστικά αυτών των αυτονόμων οχημάτων πρόκειται να αλλάξουν το επάγγελμα του μεταφορέα. Οπότε, τι, θα γίνει με τις σχετικές λειτουργίες, πώς θα ασκείται αυτό το επάγγελμα. Αν θέλετε, πέστε μας δυο λόγια πάνω σε αυτά τα ερωτήματα, γιατί στην εισήγησή σας τίποτα από αυτά δεν θίξατε. Ευχαριστούμε, λέει ο πρόεδρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, ήδη υπάρχει τεχνολογία ούτως ώστε τα αυτοκίνητα να βαδίζουν μόνο τους χωρίς να τα οδηγεί κάποιος. Όμως, εγώ από όλα αυτά τα θετικά, έχουμε και ένα σωρό ε, προβλήματα, κάποιες προκλήσεις, τι θα γίνει με τα ατυχήματα, από τα ενδεχόμενα, τι θα γίνει με θέματα ιδιωτικότητα, θέματα απασχόληση. Θα πρέπει να φροντίσουμε την οδική ασφάλεια, αυτό να είναι μια προτεραιότητα, ιδίω να προσέξουμε τους πιο ευάλωτους, δηλαδή ποδηλάτες και πεζούς. Και μέρος της εξίσωσης βέβαια είναι η διασύνδεση των οχημάτων. Θα πρέπει να μοιράζονται και πληροφορίες, τα οχήματα και αυτό αν γίνει και στα φορτηγά τότε θα έχουμε εξοικονόμηση καυσίμων, καλύτερη ε, για τους ε, οδηγούς ακόμα και θα γλιτώσουμε από τα καυσαέρια μέχρι ένα σημείο οπότε θα πρέπει να δούμε πώς αυτή η νέα τεχνολογία θα την εκμεταλλευτούμε με βιώσιμο τρόπο. Θα πρέπει να ζυγίσουμε στόχους και συμφέροντα αλλά νομίζω ότι έτσι όπως εξέστε η τεχνολογία θα πρέπει επιγόντως να θεσπίσουμε ένα νομοθετικό πλαίσιο. Και εμείς θα είμαστε στο πλάι σας, Επίτροπε. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Πώς παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η συζήτηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα βεβαίω. Και είναι απαραίτητο, κυρία Επίτροπε, να ετοιμάσει η Επιτροπή κατάλογο των ε, διαδικασιών που θα πρέπει να δοκιμαστούν σε σχέση με τα αυτόνομα αυτά αυτοκίνητα. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα που μας απασχολούν. Τα νομικά βεβαίως, οι υποδομές που πρέπει να προσαρμοστούν και η κυβερνόσφαλη για τα νομικά θα πρέπει να αλλάξει το νομικό πλαίσιο με βάση βέβαια την επικουρικότητα αλλά και θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να διαφυλαχθούν τα εθνικά χαρακτηριστικά της νομοθεσίας. Σε περίπτωση ατυχήματο επίσης, τι θα γίνει, ποιος θα έχει την ευθύνη όταν έχει προξενήσει ένα ε, αυτόνομο όχημα το ατύχημα. Ποιος θα φέρει την ευθύνη. Σε αυτό πρέπει να δώσουμε ευρωπαϊκές απαντήσεις. Και πρέπει να δώσουμε απαντήσεις και για τις υποδομές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Σάντερ. μισή λεπτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, το αυτόνομο αυτοκίνητο είναι ένα τεχνολογικό όνειρο που κοντεύει να γίνει πραγματικότητα. Σήμερα έχουμε ήμι αυτόνομα οχήματα, τα οποία παρκάρουν μόνα τους, στρίβουν μόνα τους και φρενάρουν μόνα τους. Μεθαύριο ο οδηγός θα είναι απλώς επιβάτης στο όχημά του. Κερδίζουμε χρόνο, ε, πιο αναπαυτική διαδρομή, σίγουρα. Αλλά σε επίπεδο ασφάλειας περιμένουμε μεγαλύτερη πρόοδο. Γιατί από τους 26.000 θανάτους στους ευρωπαϊκούς δρόμους οφείλονται σε ανθρώπινο σφάλμα. Πόσες ζωές θα μπορούσαμε να σώσουμε λοιπόν με την αυτή τεχνολογία. Παρ' όλα αυτά παραμένουν πολλά εμπόδια και πολλά ζητήματα σε κρεμότητα που πρέπει να λυθούν. Τα ζητήματα αυτά τα αναφέραμε. Ποιο θα είναι υπεύθυνο στην περίπτωση ατυχήματο, πώ να προσαρμόσουμε τι οδικέ μας υποδομές και τις τηλεπικοινωνίες μας ανάλογα. πώ να συντονίσουμε τη χρήση, τη δράση των διαφόρων χρηστών των δρόμων μας. Εξάλλου, τα αυτόνομα οχήματα θα είναι δίχως άλλο συνδεδεμένα. Οπότε πώς θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν hacker που θα τα κάνουν ό,τι θέλουν. Πώς λοιπόν θα αντιμετωπίσουμε συντονισμένα σε όλα αυτά τα ζητήματα. Η Ευρώπη μπορεί να έχει ηγετική θέση σε αυτήν τη νέα τεχνολογική επανάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τώρα, περνάμε στο Catch the Eye. Πρώτα απ' όλα, Ευχαριστώ. Πρόεδρε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι οι εξελίξεις προχωράνε πολύ γρήγορα όσον αφορά την αυτόνομη οδήγηση. Σε λίγο καιρό θα έχουμε μια μερικώς αυτόνομη οδήγηση, το παρκάρισμα θα γίνεται εντελώς αυτόνομα και επίσης θα υπάρχει και βοήθεια στην περίπτωση η Ευρώπη λοιπόν πρέπει να έχει μία στρατηγική για να προσαρμόσει επιγόντως την νομοθεσία της αυτή τη νέα πραγματικότητα. Όσον αφορά την ασφάλεια, όσον αφορά την νομική ασφάλεια, ακούστηκαν πολλά επιχειρήματα όσον αφορά την τυποποίηση των οχημάτων. Όντως είναι κάτι που πρέπει να γίνει πολύ σύντομα τότε σχέδια έχουμε τώρα στο μέλλον για την βελτίωση των υποδομών στις χώρες μέλη, πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτή την καινοτομία στον τομέα των οχημάτων. Ευχαριστούμε. Συν Κέλλη τώρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρόεδρε, η συζήτηση αυτή βρίσκω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Έχουμε βέβαια κάποιες ερωτήσεις. Ίσως μπορεί να απαντήσει η Επίτροπος, αλλιώς ανευθέτω όπου χρόνο. Πρώτα απ' όλα, πόσο το κοινό αποδέχεται την αυτόνομη αυτή οδήγηση. Θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος όπου θα έχουμε λίγα τέτοια οχήματα και όλο και περισσότερα όσο περνάει ο καιρός. Δεύτερον, την ευθύνη. Ποιο θα έχει την ευθύνη σε περίπτωση ατυχήματο, Ο επιβάτη, ο ιδιοκτήτη που μπορεί να μην είναι επιβάτη εκείνη τη στιγμή. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Και βέβαια το κόστος. Ξέρετε πόσο θα κοστίσουν αυτά τα οχήματα. Είναι ζωτική σημασία νομίζω και μετά το COP21 να ξέρουμε κατά πόσο θα εκπέμπουν περισσότερα ή λιγότερα αέρα του θερμοκηπίου. Ευχαριστούμε. Και πάλι ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, λέει ο κύριο Τζαμπάσκη, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που βοήθησαν να συζητήσουμε σήμερα το θέμα. Προχωράει γρήγορα τεχνολογία και η αυτόνομη οδήγηση θα πρέπει να είναι κάτι που θα πρέπει να μας ε, απασχολήσει και να είναι πρωτοπόρα στην καινοτομία η Ευρώπη είναι, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε, να προσέξουμε ε, να τηρείται η νομοθεσία που αφορά την οδήγηση. Μου λένε ότι η αυτόνομη οδήγηση θα βοηθήσει όσον αφορά την κίνηση, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο. Ευχαριστούμε. Ο επόμενος. Ξέρετε, πολλά θέματα. Τα συζητήσαμε σήμερα όσον αφορά την αυτόνομη οδήγηση. Η κυρία Επίτροπε θα πρέπει να έχει η ασφάλεια την προτεραιότητα. Αλλά έχουμε και άλλα ζητήματα να μας απασχολήσουν. Θέματα κοινωνικά, ηθικά, περιβαλλοντικά, αλλά και τεχνολογικά. Επίσης, θα πρέπει να φροντίσουμε και την προστασία των δεδομένων να δούμε πώς θα έχουμε υποδομή και ποιος θα χρηματοδοτήσει την υποδομή για τα αυτόνομα οχήματα. Τώρα, έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ευκαιρία να λάβει τον πρωταγωνιστικό ρόλο για αυτές τις εξελίξεις στην αυτοκινητοβιομηχανία και έτσι να βοηθήσετε γενικότερα την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Άρα θα πρέπει να λυθούν τέτοιες προσπάθειε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ τους πιο δραστήριους ευρωβουλευτές. Δέκατο όλων. Και τώρα, ώρα να λάβει το λόγο. Η αξιαγάπητη προσκεκλημένη μας κυρία Μαριάν Τάισεν, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ τους συναδέρφους, τους Ευρωβουλευτές για την βοήθειά τους και που παράμειναν εδώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί Ευρωβουλευτές, εδώ είμαστε αντιμέτωποι με νέα τεχνολογία, με την ανάπτυξη νέας τεχνολογίας η οποία αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα και δεν ξέρουμε από πριν, από πριν ακριβώς πού θα μας φέρει. Πολλές ερωτήσεις βέβαια έχουμε και γι' αυτό ακριβώς παρακολουθούμε και πρέπει να παρακολουθούμε την τεχνολογική εξέλιξη. Πολλές είναι οι πτυχές που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, όπως είπατε, πρέπει να υπάρξει το θέμα της ανταγωνιστικότητας, της ευθύνης, των ε, συνεπειών, της προστασίας των δεδομένων, του ιδιωτικού βίου, η χρηματοδότηση. Ποιος θα πληρώσει το κόστος για τις νέες υποδομές, τους νέους δρόμους που θα πρέπει να φτιάξουμε για να τα αποκρίνονται σε αυτήν την τεχνολογία. Θα είναι ε, κρατικά χρήματα, θα είναι ιδιωτικά, θα είναι συνδυασμό. Ε, ο κυκλοφοριακό πώς θα ρυθμίζεται, ποιος θα πληρώνει, οι χρήστες ή οι έλεγχοι, οι επιθεωρήσεις των οχημάτων, ε, νέες προδιαγραφέ ίσως για το κλίμα, με εξέλιξη όσον αφορά το κλίμα. Όλα αυτά είναι ερωτήσει που θα κληθούμε να απαντήσουμε. Η σημερινή συζήτηση ήταν χρήσιμη, αλλά είναι μόνον η πρώτη μέσα σε πολλές που θα ακολουθήσουν. Είμαστε στην αρχή, στο σημείο κίνησης ακόμα, προκειμένου να κατανοήσουμε όλες τις επιπτώσεις αυτών των νέων εξελίξεων και να τις χρησιμοποιήσουμε όσο γίνεται πιο θετικά γίνεται. Πρέπει να ξέρουμε ποιε θα είναι επιπτώσεις για τις μεταφορές και για την κοινωνία μας, το σύνολό τη, αλλά και για την ανταγωνιστική μας θέση. Έχουμε ξεκινήσει. Πράγματι, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αφήνει τα πράγματα απλώ να γίνονται. Ήδη από το 2014 έχει μία πλατφόρμα, το ξέρετε, που είναι συνεργασίας, ώστε να παρακολουθούμε όλα όσα λαμβάνουν χώρα μπήκε το πρώτο πετραδάκι θα έλεγα με την τελική έκθεση του Ιανουαρίου του 2016 και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να δημοσιεύσει ένα master plan κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά ακόμα για να παρακολουθήσει την υπόθεση αυτή. Υπάρχει και η ομάδα υψηλού επίπεδου για την αυτόνομη οδήγηση που παρακολουθεί τις εξελίξεις για να υπάρξει ένας χάρτης πορείας. Στα πλαίσια του GR33 επίσης υπάρχει διαβούλευση όσον αφορά την αυτόνομη οδήγηση. Όλοι μαζί λοιπόν, και γι' αυτό και η Επιτροπή θα ετοιμάσει το Master Plan, ελπίζουμε ότι θα έχουμε ένα σχέδιο φέτος για να καταλήξουμε σε μια πράσινη βίβλο την οποία σίγουρα θα σας παρουσιάσουμε εδώ και ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία πολλές φορές ακόμα να καθίσουμε και να συζητήσουμε με τους 10 ή με παραπάνω ίσως γι' αυτό το τόσο σημαντικό ζήτημα προκειμένου να το παρακολουθήσουμε. Ας ευχηθούμε καλή συνεργασία και καλή κατάληξη. Πολλές είναι οι εξελίξεις, ας τις αντιμετωπίσουμε θετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Επίτροπε για την παρουσία σας εδώ και για τόσο μας είπατε. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους ευρωβουλευτές που παρέμειναν στην αίθουσα και για τα πολύτιμα σχόλιά τους. Είμαστε λίγοι, αλλά σίγουρα οι καλοί. Οπότε, κυρίσω τη λήξη της ε, συζήτησης καταρχήν.